αν και ο κίνδυνος για να κολλήσουν την ασθένεια ε, αυτοί που συνταξιδεύουν θεωρείται ε, πάρα πολύ χαμηλός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το Συμβούλιο λοιπόν. Έχει κλείσει η συζήτηση. Πριν περάσουμε στην επόμενη συνάντηση θα ήθελα να κλείσουμε το θέμα των πρακτικών στα γαλλικά. Εγώ ζήτησα να ελέγξουν οι υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου την εφαρμογή του κανονισμού σε σχέση με τις τροπολογίες. Το άρθρο 192 λέγει στο σημείο του 3 εφόσον τα πρακτικά αμφισβητηθούν τότε το Κοινοβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίζει για το αν θα ληφθούν υπόψη οι αλλαγές οι οποίες έχουν ζητηθεί κανένας βουλευτής δεν μπορεί να πάρει το λόγο για πάνω από ένα λεπτό. Είχα ζητήσει λοιπόν κύριε Γκόλνης, ποια είναι η τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε. Ε, σας σέβομαι κύριε Γκόλνης και γι' αυτό ακριβώς σας απαντώ. Σας απέστειλα την τελική απάντηση γιατί θα ήθελα να σας δώσω εγγυήσει για, για τον ρόλο σας ως βουλευτή. Λοιπόν, είχα δίκιο, το έλεγξα όπως σας είπα και σας ζητώ, εάν υπάρχει τώρα μία τροπολογία από δική σας πλευράς, δεν μιλάμε για πολιτικές τροπολογίες, δεν κάνουμε μία πολιτική συζήτηση. Εάν υπάρχουν λάθη επί του κειμένου, μπορείτε να προτείνετε τροπολογίες. Άλλος πώς θα απορρίψω την τροπολογία σας, γιατί όπως σας είπα, το κείμενο αυτό λέγει ότι μόνο στην περίπτωση που χρειάζεται θα υπάρξει αλλαγή. Υπάρχει λοιπόν μία τροπολογία. Είναι αποδεκτή η τροπολογία. Αν όχι, τότε γίνεται δεκτό το κείμενο ως έχει. Ο κύριος Γκιόλνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που προχωράτε στην ψηφοφορία αυτή. Δεν είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός γιατί η παράγραφος 2 ομιλεί για έγκριση ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει την απόρριψή του του σημείου 6. Θέλετε να προχωρήσετε μέσω τροπολογίας. Προτείνω την εξή λοιπόν, η οποία συμπληρώνει την πρώτη παράγραφο του άρθρου 6 των πρακτικών. Λοιπόν, έχει ως εξή η τροπολογία μου. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών ε, ε, γίνεται η ψηφοφορία ταυτόχρονα και σε σύνδεση με τη Χόβνα Ράντα της Ουκρανίας. Και η τροπολογία μου λέει το εξής. Η φράση είναι η εξής. Η μη κανονική αυτή διαδικασία, ιδιαίτερος έκτακτη, δεν τέθηκε στην έγκριση των Ευρωπαίων Βουλευτών. Πρόκειται για μια μη τακτική και ευνίδια διαδικασία η οποία δεν τέθηκε προς έγκριση από τους ευρωβουλευτές. Αυτά. Νομίζω ότι έτσι συμπληρώνουμε τα πρακτικά με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να λέγουμε ακριβώς τι κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Κύριε Γκόλνης, δέχομαι τις ιδέες σας όπως πάντα. Δέχομαι και σέβομαι τις ιδέες σας. Αλλά η τροπολογία σας είναι ένα πολιτικό σχόλιο σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβη. Δεν υπήρξε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σχόλιο επί αυτών τα οποία συνέβησαν. Λοιπόν, η τροπολογία δεν είναι αποδεκτή. Τελείωσε. Δεν, δεν θα συνεχίσουμε. Έκλεισε το θέμα. Θα συνεχίσουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε τη δήλωση της α, α, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάτης εκπροσώπου της Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ, την κατάσταση στη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ίσης περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων.